Θα εξετάσουμε τώρα την έκθεση της κυρίας Πόλσεν για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων από το 2012 μέχρι και το 2015. Να δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διατύπωση αυτής τη στρατηγικής για την καλή διαφύωση των ε, ζώων με απασχόληση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και για οι σκιώδεις συζητητές υπήρξαν εξαιρετικοί. Καταφέραμε να επιτύχουμε μια συμφωνία επί όλων των θεμάτων. Συμφώνησαν οι οργανώσεις, οι γεωργοί, αλλά παρέμειναν ορισμένα βασικά σημεία, ορισμένα ευαίσθητα σημεία. Ένα από αυτά φορά νομικά θέματα. Θεωρήσαμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις χώρες μέλη κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περίοδου. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που συνέβη με τους ε, κλωβούς των ήθων. Υπήρξε μια περίπτωση, μια περίοδος τεσσάρων ετών κατά τη διάρκεια του, της οποίας ε, δεν μπόρεσε η Επιτροπή να κάνει τίποτα. Θα πρέπει να Έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να ελέγχουμε, θα πρέπει πάντοτε η κάθε χώρα μέλος να λογοδοτεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία συμπεριλαμβάνει μια μεταβατική περίοδο. Το νομικό πλαίσιο εδώ είναι κάπως αμφιλεγόμενο. Ένα άλλο αμφιλεγόμενο θέμα για το οποίο διεξήχθη μια εκτενή συζήτηση αφορούσε την σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα πρέπει να ε, μπαίνει μια σήμανση στο κρέας. Προσωπικά βρίσκω ότι είναι λάθος αυτό. Καταρχάς, θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον ε, δεν υπάρχει μια κατάχρηση ορισμένων εξαιρέσεων θρησκευτικού χαρακτήρα. Γιατί πιστεύω ότι όποιος παρεκκλίνει ή όποιος καταχράται αυτή την εξαίρεση δεν θα γράψει ποτέ πάνω, δεν θα βάλει σήμανση ότι η σφαγή δεν έγινε με αναισθητοποίηση. Το τρίτο σημείο αφορά τα stray dogs, οι stray cats, δηλαδή τα 20 τα ζώα που γίνονται αδέσποτα. Ναι. Στο έγγραφό μας αποδίδουμε μεγάλη σημασία, στις ε, δίνουμε την ευθύνη στις μεμονωμένες χώρες μέλη και στις τοπικές οργανώσεις ό,τι αφορά τα δέσποτα ζώα. Ε, εκφράζουμε την επιθυμία όλα τα τα ζώα να φέρουν ένα διακριτικό. Αυτό που είναι σημαντικό όμως σε αυτή την πρόταση είναι να υπάρξει μια γενική νομοθεσία για την προστασία των ζώων συγκρίσιμη με αυτή που ισχύει για τα τρόφιμα. Μία νομοθεσία η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ζώα με εξαίρεση τα άγρια. Μια στρατηγική η οποία θα έχει σαφείς ορισμούς ως προς τη σημασία που έχει μια προσεκτική φροντίδα των ζώων. Μια νομοθεσία η οποία θα καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Εκτός από αυτό θα πρέπει να ε, διαδοθούν και ορισμένα στοιχεία για τα θέματα αυτά. για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις ε, ε, διάφορες προτάσεις ε, που έχουν γίνει. Ας μην ξεχνάμε την, την κλωνοποίηση. Ξέρουμε ότι μετά από την κλωνοποίηση η ζωή δεν μπορεί να είναι φυσιολογική. Οι γενικοί κανόνες επιτρέπουν τον ίσο ανταγωνισμό για όλους τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Πασάσκου. Το θέμα που συζητήσαμε σήμερα συζητάμε βασικά το θέμα των ζώων συντροφιά και των οικόσιτων ζώων. Θα ήθελα όμω να μιλήσω για τα δελφίνια στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί κινδυνεύουν. Πάνω από 300 δελφίνια πέρασαν στη Μαύρη Θάλασσα τα τελευταί, τους τελευταίους μήνες. Είναι θύματα παράνομης αλληλείας και πραγματικά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι μπροστά στο δράμα που βιώνουν αυτά τα όμορφα και έξυπνα ζώα. Για το λόγο αυτό υποβάλαμε μια γραπτή δήλωση την υπαριθμών 24. Ζητάμε να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να προστατεύσουμε αυτά τα, τα, τα ζώα χρησιμοποιώντας εξοπλισμούς ήχου. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να υπογράψουν την δήλωση αυτή για τα δελφίνια. Οι καταναλωτές ε, περιμένουν ότι τα ζώα στα, ε, στις εκμεταλλεύσεις ε, θα αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρονται. Ε, είναι πολύ σημαντικό να είναι σωστά τα πρότυπα για την καλή υγεία των ζώων και επηρεάζουν όλο και περισσότερο και το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που τους δίνει το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου της Ένωσης και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 ώστε να προωθήσουν την εφαρμοσμένη έρευνα στην καλή κατάσταση των ζώων και να βρουν και καινοτόμες λύσεις για την καλή υγεία και καλή κατάσταση των ζώων. Πάνω σε αυτή τη βάση πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επενδύσουν πιο πολύ στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την υγεία των ζώων. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ταμπάτζη. Ευχαριστώ κύριε. κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, μιλήσατε για την ε, Ουγγαρία και για τις ε, παραγωγούς όνειρες, υπήρξε μια παρεξήγηση. Πιστεύω ότι πιστεύουν πολλοί ότι αυτό είναι κάτι που εφίδραν οι γραφειοκράτες της, ε, των Βρυξελών, άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ με μια ζωντανή όρνηθα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο κανονισμός αυτός είναι πολύ οπισθοδρομικός. Όλες οι χώρες ε, μέλη είχαν ε, ε, αρκετά χρόνια για να μπορέσουν να συμμορφωθούν και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις ε, σε ό,τι αφορά τις όνειθες. Δυστυχώς υπήρξαν διπλά πρότυπα μεταξύ των χωρών μελών. Συνεπώς ε, δεν καταφέραμε να αυξήσουμε το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά μείναμε έκπληκτοι μπροστά σε αυτά τα μέτρα Έχετε το λόγο. Ε, μπλε κάρτα στον κύριο Ταμπάτζη. Ε, Συγγνώμη που χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο της μπλε κάρτας. Ήθελα μόνο να πω ότι θέλω να συμμετάσχω και να πάρω το λόγο. Καλώς. Να δώσω τότε το λόγο στην κυρία Λιωτάχ. Κοιτάξτε, η στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων έχει ενδιαφέρον, όμως πολλά ζώα δεν συμπεριλαμβάνονται σε την πρόταση αυτή. Σε ένα άλλο ψήφισμα είχα προσθέσει δύο σημεία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ε, υπέρ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλούμε για το περιορισμό της διάρκειας του χρόνου μεταφοράς μέχρι τα σφαγεία. Δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η διάρκεια αυτή και πολλοί έχουν υπογράψει αυτή την αναφορά. Η πλειονότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει πιο βραχία διάρκεια στην μεταφορά μέχρι το σφαγείο. Από εκεί και πέρα έχουμε και την απαγόρευση των προϊόντων ε, κλωνοποίησης, των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων και όλων αυτών. στην ε, μεγαλύτερη πλειοψηφία ε, τα νεκρά ζώα είναι το αποτέλεσμα της ε, κλωνοποίησης και δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι η τελευταία ευκαιρία για να κάνουμε μια χειρονομία προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κυρία Λιωτάχο, κύριος Βοσισόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Πόλσεν για την εξαιρετική της έκθεση έχετε εξετάσει το θέμα αυτό με ρεαλισμό και με ευαισθησία, συνάμα. Οι προτάσεις σας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και οι προτάσεις σας είναι πολύ σωστά τεκμεριωμένες. Ωστόσο, ως προς τη χρηματοδότηση, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την καλή διαβίωση των ζώων χωρίς επιπρόσθετη βοήθεια ή χρηματοδότηση. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, μεγάλο μέρος της ε, έκθεσής σας το αφιερώνεται ε, στο εμπορικό σκέλος ε, και στη θέση που θα πρέπει να έχει η καλή διαβίωση των ζώων στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να απαιτούμε τις προϋποθέσεις αυτές να τις σέβονται και όσοι εισάγουν ε, ε, ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει ο κύριος Σκότα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάριν Πούλσερ για την έκθεση μου φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος που λόγω ενός αναχρονιστικού πνεύματος μας κάνει να χάνουμε χρόνο και αυτό έχει ανετικές επιπτώσεις σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Μπροστά σε ένα κείμενο που παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους φίλους των ζώων, όπου συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, που έχει θετικές επιπτώσεις στα ίδια τα ζώα, θέλουμε να προτείνουμε τροπολογίες οι οποίες στρεβλώνουν όλη την σημασία της ε, καλής διαβίωσης με ασαφείς προτάσεις. Συνεπώς δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ αν θα πρέπει να επενδύσουμε χρόνο και πόρους για να εξετάσουμε προτάσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες. Συνεπώς θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης κυρίας Πούτσεν. Ο κύριος Πάσκα είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η δυσκολία στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δημιούργησε για πάρα πολύ καιρό το περιθώριο για απάτες. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η οδηγία για τις οτοπαραγωγούς όρνηθες. Για 12 χρόνια χρησιμοποιήθηκαν τα καινούργια αυτά κλουβιά και σε κάθε περίπτωση δεν είναι έτοιμες όλες οι χώρες για να τις Η Ουγγαρία, η Πολωνία, παρα... Ε, αναβάλουν συνέχεια τη χρήση και αναρωτιόμαστε αν είναι έτοιμες να ετοιμάσουν τους κλοβούς αυτούς για τις οπαραγωγούς όρνηθες. Τι συμβαίνει με τα αυγά που προέρχονται από αυτές τις όρνηθες. Ε, υπήρξε ένα σκάνδαλο τον περασμένο Ιούνιο στην ε, Σλοβακία γιατί ξέσπασε μία επιδημία σαλμονέλωσης. Αρρώστησαν 56 παιδιά και οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι υπήρχαν αυγά που προερχόντουσαν από χώρες με ε, ε, ψευδείς Δίνουμε τώρα το λόγο στον Επίτροπο Νταλή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές εκδηλώσεις και συζητήσεις έγιναν φέτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και αλλού στο φως της ανακοίνωσης της Κομισιόν που παρουσίασε την ε, στρατηγική της Ένωσης για την καλή διαβίωση, διαβίωση των ζώων, η οποία στρατηγική προτείνει μια νέα προσέγγιση για το μέλλον της ε, καλής διαβίωσης των ζώων στην Ευρώπη. Μετά από περίπου 40 χρόνια νομοθεσίας υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωση σε αυτό το τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική αφορά την καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης, καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο, επικέντρωση στην εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη στους εμπλεκομένους σε επίπεδο βάσης. Πριν μπω σε επιμέρους θέματα, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το εξαιρετικό έργο της εισηγήτριας κυρίας Πάουλσεν, η οποία παρουσίασε ισορροπημένη έκθεση σε αυτό το σύνθετο και πολύ ευαίσθητο τομέα. Ε, χαίρομαι που σημειώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις απόψεις της Κομισιόν για τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής. Ε, πρόταση απλουστευμένου νόμου πλαισίου που λαμβάνει υπόψη επιμέρους ιδιαιτερότητες ε, ειδών και τομέων, καλύπτει όμως όλα τα ζώα ε, στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κέντρων αναφοράς για την καλή υγεία των ζώων για να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές θα παίρνουν την ίδια τεχνική πληροφόρηση σχετικά με το πώς θα εφαρμόζονται οι νομοθεσίες της Ένωσης και να διαδίδουν ε, τεχνογνωσία, πορίσματα έρευνας, τεχνικές καινοτομίες Ανάπτυξη δικτών για την καλή διαβίωση των ζώων στο νόμο πλαίσιο για να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα για την καλή τους διαβίωση και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα ε, πρακτικής φύσεως που πρέπει να ληφθούν υπόψη και ε, εισαγωγή νομικών οροσίμων ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη νέα νομοθεσία. Επίσης η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίσουμε καλύτερη επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας και αυτό είναι κεντρική σημασία για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμερίζομαι επίση απόψει που εκφράστηκαν στην έκθεση τη κυρία Πάουλσεν σχετικά με τη σημασία υποστήριξη και βελτιστοποίηση τη διεθνού συνεργασία στην ε, πολυμερή αρένα παγκοσμίως ιδιαίτερα των ΦΑΟ και τον, ε, την, Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων ε, και σε διμερείς διαπραγματεύσεις ε, που βάζουν το θέμα της καλής διαβίωσης των ζώων στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και την προώθηση των απόψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανόηση των προτύπων. Ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό επειδή η παραγωγή των τροφίμων έχει γίνει παγκόσμια δραστηριότητα που επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία της έκθεσης στα οποία επί των οποίων η Κομισιόν δεν έχει ακόμα αποφανθεί οριστικά και νομίζω ότι η περισσότερη σκέψη χρειάζεται πριν προτείνουμε ε, πιθανές δράσεις. Ε, για παράδειγμα, η έκθεση προτείνει η Κομισιόν να εξετάσει, να αναπτύξει ένα συνεκτικό ε, πρόγραμμα σήμανσης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους παραγωγούς που θα ξεπερνάει την τωρινή νομοθεσία για την, ε, την σήμανση. Και εγώ θα ήθελα οι παραγωγοί της Ένωσης που επιθυμούν να βελτιώσουν την καλή διαβίωση να έχουν καλύτερη τιμή για τα ζώα τους θα πρέπει όμως να το εξετάσουμε αυτό. Επίσης ε, η έκθεση ζητάει υποχρεωτικά μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Όπως θα ξέρουν τα αξιότιμα μέλη, η αναθεώρηση του κανονισμού για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου είναι κομμάτι της αναθεώρησης της ΚΑΠ. Αυτή η ιδέα λοιπόν θα εξερευνηθεί καλύτερα μέσα στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Όμως ημερίζομαι την άποψη που εκφράζει ο εισηγητής σχετικά με τη βελτίωση της συνοχής, της συνεκτικότητας στη συνολική προσέγγιση. Η καλή διαβίωση των ζώων είναι ένα οριζόντιο θέμα και πολλές πολιτικές επηρεάζονται. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να θεωρήσουμε αυτή την πρόταση πάρα πολύ χρήσιμη και σωστή. Ας δούμε τώρα τα ζώα συντροφιάς. Η Κομισιόν έχει συμφωνήσει να κάνει μια σειρά μελετών συμπεριλαμβάνοντας και το συγκεκριμένο θέμα στα πλαίσια της στρατηγικής και πάνω στη βάση των αποτελεσμάτων αυτού του εγχειρήματος θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάμε παραπέρα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι η μεταφορά των ζώων και έχει να κάνει με την καλή διαβίωσή τους. Είχα τη χαρά και την τιμή να δεχθώ μια αντιπροσωπεία πριν από μια ε, εβδομάδα ε, που είναι υπεύθυνη για τα όρια της μεταφοράς και είχα την ευκαιρία να εξηγήσω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα αιτήματα μείωσης των αποστάσεων για δύο λόγους και θα δούμε το θέμα στα πλαίσια της αναθεώρησης του βασικού νόμου για την καλή διαβίωση των ε, ζώων που είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής που συζητάμε. Και προτείνουμε μεταξύ άλλων νέα εργαλεία για την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας ε, συμπεριλαμβανομένης ε, και της διάρκειας της μεταφοράς. Πρέπει να πω ότι η επιβολή είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η Κομισιόν δεν θα κάνει ε, αλλαγές στον κανονισμό για τη μεταφορά. Στο Συμβούλιο 18 Ιουνίου είπα ότι προτείναμε ευρία γκάμα δράσεων νομοθετικών και άλλων για να βελτιώσουμε στις την καλή διαβίωση στη μεταφορά. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, το θέμα των μακρών αποστάσεων ε, που πρέπει να καλύψουν τα ζώα μέχρι το σφαγείο. Είμαι έτοιμος να εξετάσω όλα τα δεδομένα τα οποία θα φωτίσουν το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τις προτινόμενες δράσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την καλή διαβίωση, τις δράσεις που προτείνονται, γιατί υπάρχουν πολλές δράσεις που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά. Ε, ορισμένα άλλα θέματα για τις παραγωγούς ορνηθές και τις κλωβούς, ε, τους κλωβούς πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια οδηγία που θεσπίστηκε πριν από 12 χρόνια στο τέλος της μεταβατικής περίοδου ε, μέχρι το τέλος του περσινής χρονιάς και το γεγονός ότι κάποιες χώρες είχαν βραχύτερο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν και να αλλάξουν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή οι χώρες αυτές και η δική μου είναι ανάμεσα σε αυτές διαπραγματεύτηκαν την οδηγία αυτή κατά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Οπότε δεν ήταν απόλυτα σαφές ποιος θα ήταν ο χρονικός ορίζοντας και οι δεσμεύσεις. Για την κλωνοποίηση πολλές φορές ε, έχω πει ότι τώρα η Κομισιόν διεξάγει μία εις βάθος ε, ανάλυση επιπτώσεων στο θέμα αυτό της κλωνοποίησης και κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με πρόταση για μια οδηγία ανεξάρτητη για την κλωνοποίηση. Ε, να ευχαριστήσω πάλι το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την κυρία Πάουλσεν και την ομάδα της για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Προσβλέπω ε, στην περαιτέρω πρόοδο από κοινού, από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, ε, καθώς θα εκτιλήσετε τη στρατηγική μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρών τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε επί του κειμένου την Δετάρτη στις 12.30. Ξεκινούμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση Κοχ και Σενάλ.